δεν μπορώ να παραμείνω σε αυτή τη θέση και να στηρίζω αυτή την απερίσκεπτη θεωρώ προσέγγιση όσον αφορά τη μελλοντική εργασία των αντιπροσωπιών μας. Σας ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Λυπούμε για αυτό το οποίο κάνετε. Βεβαίως ε, Πράγματι είχατε συντάξει και μια σχετική επιστολή όσον αφορά την ομόφωνη απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Λυπούμε λοιπόν, αλλά βεβαίως δεν μπορώ να αλλάξω την απόφασή σας. Κυρίες και κύριοι, πριν ε, περάσουμε στην ε, ψηφοφορία της έκθεσης Φερέρα για την Τραπεζική Ένωση, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση και να πω ορισμένα πράγματα προς κάποιους συναδέλφους. Όλοι ξέρουμε πως η Τραπεζική Ένωση είναι οπωσδήποτε ένα ιστορικό βήμα και νομίζω πως ε, είναι, αν εγκριθεί τώρα στην ε, ψηφοφορία, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτής της ε, θητείας μας. Είναι οπωσδήποτε ιστορικό και συγκρίνεται μόνο με την εσωτερική αγορά το Κοινοβούλιο Βεβαίω εργάστηκε πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό οφείλω εγώ ως ε, πρόεδρος ε, να πω πως έπρεπε να σπάσει αυτή η σύνδεση μεταξύ των ε, τοξικών χρεών των τραπεζών και θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω πολλούς συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πέντε γυναίκες και ένας άνδρας ε, που πάλεψαν πραγματικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά την Ελίζα Φερέρα, την Κορίν Βόρτμαν Κόλ, την Σάρον Μπόουλς, την Σιλβί Γκουλάρ, την Βικτόρια Φόρτ και τον Σβεν Γκίγκολντ που πραγματικά έφτασαν στα όρια της φυσικής τους αντοχής παλεύοντας για τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Οπωσδήποτε ο καθένας αξιολογεί διαφορετικά το τελικό αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ εγώ πως ε, ήταν εξαιρετικό και οπωσδήποτε υποδειγματικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματευτήκατε. Πριν από την ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Φερέρα, τον λόγο έχει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο κύριος Βενιζέλος. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν την ψηφοφορία να κάνω εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη δήλωση.